Okay, Συναδελφοί, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Έχουμε αργήσει λίγο. Θα ξεκινήσουμε από το σημείο 2 της ημερησίας διάταξης, διότι το πρώτο ήταν η συνεδρίαση των συντονιστών. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το σημείο 2, έγκριση της ημερησίας διάταξης. να σας ενημερώσω ότι αργότερα σήμερα θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με το ελεγκτικό συνέδριο και θα έχουμε εδώ και τον ε, κύριο Πίνγκστεν, ε, τον πρίτανη του ε, ελεγκτικού συνεδρίου και επίσης τον Κλάους Χάινερ Λίνε που είναι πρώην συνάδελφός μας. Ήθελα λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με το ελεγκτικό συνεδρίο και αύριο θα ε, έχουμε ε, προσκεκλημένους ε, κύριο Μπέκη που θα μιλήσει για τις παράνομες ροές κεφαλαίων και τον Έρικ Σόλχαμ από το ΟΣΑ. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε αθρώα προσέλευση ευρωβουλευτών. Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημείο 3. Ανακοινώσει ε, της Προέδρου. Μία ανακοίνωση έχω που έχει να κάνει με τον Μπουρούντι, διότι υπήρξαν εξελίξεις εντός του Συμβουλίου πάνω στο θέμα του Μπουρούντι. Πριν ένα χρόνο περίπου ήμουνα στο Μπουρούντι με τον ε, πρόεδρο της ε, Ομάδα των σοσιαλιστών ε, και τότε φαίνονταν αρκετά ήσυχα τα πράγματα και είναι ε, φρικτό να σκέφτεται κανείς τι συμβαίνει ε, εκεί τώρα. Στις 14 Μαρτίου το Συμβούλιο ολοκλήρωσε τις διαβουλεύσεις με τον Μπουρούντι σύμφωνα με το άρθρο 96 της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ, της Συμφωνίας Κοτονού οι δεσμεύσει ε, τη ε, κυβέρνηση ε, του Μπουρούντι δεν ακούνε για να καλύψουν τι ανησυχίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναστείλει την οικονομική της βοήθεια προς την κυβέρνηση. Συνεχίζει όμως την χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπάρχουν θέματα με, το, με τη Ρουάντα, ε, υπάρχουν ενισχυτικές εξελίξεις στην περιοχή των μεγάλων λιμνών. Και ε, αυτό το μήνα ε, έχουμε την 22η επέτειο της γενοκτονίας της, των Τούτσι στην Ρουάντα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Ελπίζουμε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στην περιοχή. Απλά ήθελα να σας πω ότι έχουμε να στείλει την οικονομική βοήθεια προς την κυβέρνηση του Μπουρούντι. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης σε πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης ε, της 17 7η και 18 η Φεβρουαρίου και τη 14 η και 15 η Μαρτίου. Βρίσκονται στο φάκελό σας. Εάν έχετε παρατηρήσει, σας παρακαλώ ενημέρωση τη γραμματεία πριν το τέλος ε, της συνεδρίασης. Εάν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, θα θεωρηθεί ότι εγκρίθηκαν τα πρακτικά. Σημείο 5 της ημερησίας διάταξης, έγκριση αποφάσεων και συστάσεων των συντονιστών ε, ε, της ε, συνεδρίασης της 16ης Μαρτίου. Και πάλι, αν έχετε παρατηρήσει, σας παρακαλώ ενημερώστε μας μέχρι το τέλος ε, της συνεδρίασης. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θα θεωρηθεί ότι εγκρίθηκαν. Σημείο 6, ανακοινώσει της Επιτροπής. Δεν ξέρω ποιος εκπρόσωπος της Επιτροπής βρίσκεται εδώ. Δεν έχουμε ανακοινώσει από την Επιτροπή. Πολύ ωραία. Αργότερα σήμερα θα έρθει ο Επίτροπος Στυλιανίδης θα μπορέσει λοιπόν εκείνο να μα ενημερώσει. Σα ευχαριστώ πολύ. Α, ακριβώς στην ώρα του ε, βλέπω ότι ε, καταφτάνει ο εισηγητή του σημείου 7. Το σημείο 7 λοιπόν είναι η γνωμοδότησή μα προ την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγή για του σκοπού κοινών διαδικασιών που αφορούν τη χορήγηση και ανάκτηση του καθεστώτο διεθνού προστασία. Έχει να κάνει με το άσυλο δηλαδή το θέμα αυτό. Η ΛΥΜΠΕ είναι αρμόδια επί της ουσίας. Ε, θα ψηφίσουμε την ε, γνωμοδότηση σήμερα το απόγευμα. Ε, ο ΣΕΜΠ λέει ότι το θέμα αυτό είναι αρκετά επίμαχο. Θα πρέπει να επιλύσουμε το θέμα της κρίσης των προσφύγων. Σου δίνω λοιπόν τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας και όπως είπατε είναι πράγματι επίμαχο το θέμα αυτό είναι ένα θέμα που συνδυάζει την ε, ανάγκη μας για αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού και γι' αυτό είναι και πιο επίμαχο θέμα. Είμαι ευγνώμων προς όλους τους συναδέρφους που συνέβαλαν ε, στην έκθεση αυτή. του ευχαριστώ για τη δουλειά και υποστήριξή τους. Χαίρομαι που ως Επιτροπή μπορέσαμε να είμαστε ενωμένοι όσον αφορά το θέμα του καταλόγου ασφαλών χωρών. Το θέμα αυτό δεν είναι η ιδιαίτερη αρμοδιότητα της ΔΕΒΕ. Προτείνω λοιπόν να περιμένουμε το αποτέλεσμα της μελέτης αντικτύπου του της υπηρεσίας ε, ε, θεμελιωτών δικαιωμάτων. Ε, τώρα λοιπόν έχουμε την γνωμοδότηση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Βλέπω λοιπόν ότι χρειάζεται περαιτέρω εξέταση το θέμα αυτό. Κάτι που υποστηρίζει τη θέση της Επιτροπής μας. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που δείχνουν κάποιες ελαφρές διαφορές απόψεων μεταξύ των ομάδων. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι η Επιτροπή μας μπόρεσε για άλλη μια φορά να υιοθετήσει κοινή προσέγγιση και το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι Ε, η γρήγορη διεκπαιρέωση των ε, αιτήσεων ασύλου δεν θα πρέπει να έχει προτεραιότητα απέναντι στην προστασία των δικαιωμάτων μειονοτήτων. Χρειάζεται λοιπόν ε, η πρόταση αυτή περισσότερη εις βάθος εξέταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να ανήκει σε αυτούς που λαμβάνουν βιαστικές αποφάσεις όσον αφορά τα θέματα των προσφύγων. Χαίρομαι που ε, δόθηκε η γνωμοδότηση αυτή στην Επιτροπή μας ε, και είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται σε όλους τους τομείς που μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση του θέματος αυτού. Ελπίζω η γνωμοδότησή μας ε, να μην θεωρηθεί ότι αντίκειται στις εργασίες της Κομισιόν, αλλά, εν πάση έχουμε υποβάλει τη θέση μας. Αυτά από μένα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή ο κατάλογος ασφαλών χωρών ε, δεν συμπεριλαμβάνει αναπτυσσόμενες χώρες. Μιλάμε κυρίως για τις χώρες ε, της ε, πρώην Ιουκοσλαβίας, τη Βοσνία και την Τουρκία. Αλλά συζητήθηκε η επέκταση του καταλόγου. Ωραία, Σεπ, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σου. Θα ακούσουμε τώρα τους σκιώδεις εισηγητές. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο Μπόγκταν Βέντα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για όλη αυτή την προετοιμασία. Έχω κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά δύο τροπολογίες, την 2 και την 10. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το να μπει μια χώρα στον κατάλογο ασφαλούς, ασφαλών ε, χωρών καταγωγής δεν σημαίνει ότι υπάρχει απαραίτητα και ασφάλεια και προστασία για τους πολίτες. Θέλω να πω ότι πρέπει να ελέγχουμε στην πράξη κατά πόσο ισχύει η διεθνής προστασία. Έχω και κάποια τροπολογία για τις ε, μειονότητες, όπως για παράδειγμα η ΛΟΑΔΜΑ και άλλες ευάλωτες ομάδες. Για το 29 και 30 πρέπει να υπάρχουν εγγύησει ώστε να μην γίνονται διακρίσεις εξαιτία είτε σεξουαλικής ταυτότητας, είτε φίλου, είτε οτιδήποτε άλλο. Που να λέει ότι στην περίπτωση που οι ετούντες χρειάζονται ιδιαίτερες εγγύησεις, και δεν ε, τους προσφέρονται αυτές οι εγγύησεις, οι ετούντες αυτοί να μην ακολουθούν την συνήθη διαδικασία, αλλά να εξαιρούνται από αυτήν. Συζητήσαμε με συναδέλφους από τη ΛΥΜΠΕ για την τροπολογία αυτή και αυτοί πιστεύουν ότι καλύπτεται από την οδηγία αυτό το θέμα, ότι δεν είναι αναγκαίο. Αποκλείονται και άλλες μειονότητες, εθνοτικές ή θρησκευτικέ δεν ε, περιλαμβάνονται στην τροπολογία. Οπότε, εδώ υπάρχει έλλειψη συνοχής κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να απορριφθούν αυτές οι τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Μαρίνα Αλβιόλτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το έργο του. Ξέρετε ότι η Γκουε δεν έχει υποβάλει τροπολογία στην έκθεση αυτή, γιατί εμείς δεν συμφωνούμε με την κατάρτιση ενός καταλόγου ασφαλών χωρών. Είμαστε κατά, δηλαδή, του ίδιου του στόχου, του πνεύματος. Οπότε δεν υποβάλαμε καμία τροπολογία. Εμείς πιστεύουμε ότι η εκπόνηση τέτοιου καταλόγου ασφαλών χωρών σημαίνει ότι συνεχίζουμε με τις πολιτικές μας όπου τα σύνορά μας προστατεύονται απ' έξω και γίνονται διακρίσεις σε βάρος των μεταναστών, μεταναστριών και προσφύγων. Είδαμε τι σημαίνει να υπάρχει κατάλογος ασφαλών χωρών. Έχουμε βάλει την Τουρκία μέσα. Είδαμε τι σημαίνει η συμφωνία αυτή Ευρωπαϊκής Ένωσης με Τουρκία που οδήγησε σε βία μεταφορά και μετατόπιση του κόσμου με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο οι ζωές πολλών μεταναστών και προσφύγων. Είμαστε κατά λοιπόν της ιδέας αυτής. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. χαρτάλα. Τώρα, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ακολουθεί τη σωστή στρατηγική ο εισηγητής εδώ. όσον αφορά τις επικρίσεις για τη δημιουργία ενός τέτοιου καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής. Θέλω λοιπόν να τον ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του. Νομίζω ότι η ποιότητα της γνωμοδότησης αυτής φαίνεται και από το γεγονός ότι υπάρχουν μόνο πέντε τροπολογίες. Μία από αυτές έρχεται από τη δικιά μου ομάδα, όπου ζητάμε να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε διόρθωση, σε αποκατάσταση. Το βασικό εδώ είναι ότι το δικαίωμα στο άσυλο θα το εγγυούμαστε εν πάση περιπτώσει, και ότι οι ετούντες θα έχουν την ευκαιρία να προσβάλλει την ιδέα αυτή της ασφαλούς χώρας αν ο ίδιος προσωπικά πλήτεται για κάποιο λόγο. Είναι σημαντικό επίσης οι ετούντες να έχουν το δικαίωμα στην αποκατάσταση εφόσον υπάρξει αρνητική απάντηση. Νομίζω ότι είναι διατεθειμένος να δεχτεί την τροπολογία μας ο εισηγητής. Όλα λοιπόν αναφέρονται καλά στην έκθεση αυτή και αποτελεί ένα καλό εργαλείο και βοήθημα για την ΛΥΜΠΕ να καταλήξει στην τελική της απόφαση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Γκέρενς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση στη διαδικασία άλλη διαδικασία που εφαρμόζεται στις χώρες μας για την υποδοχή των ετούντων άσυλο και άλλο η αρχή της ασφαλούς χώρας. Δεν υπάρχει καμία χώρα απολύτως ασφαλής, εκτός ίσως αυτές που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης, παρόλο που δεν είμαι σίγουρος. Αν κάποιος έρθει στις χώρες μας, έχει δικαίωμα σε ατομική διαδικασία. Και η ατομική διαδικασία υπάρχει ακριβώς για λόγους νομικής ασφάλειας και είναι ένα μέτρο το οποίο προστατεύει νομικά και βοηθάει τον ετούντα άσυλο να ξέρει τι τον περιμένει. Δεν υπάρχει συλλογική διαδικασία εκτός αν υπάρχει ανωτέρα βία. Αλλά και πάλι ε, μετά οι ετούντες άσυλο πρέπει να περάσουν από μία εξατομικευμένη διαδικασία. Αυτή είναι η πρακτική στις χώρες μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να την αφισβητήσουμε αυτή την αρχή και να την αλλάξουμε. Δεύτερον, καταλαβαίνω πολύ καλά ότι θέλουμε εδώ να υπάρχει μια τροπολογία για να επιστήσουμε την προσοχή όλων στα άτομα ΛΟΕΔΜ αυτοί που διώκονται λόγω της σεξουαλικής τους προτίμησης έχουν δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο στις χώρες μας. Αυτό που με ενοχλεί εμένα δεν είναι η αρχή αυτή. Είναι το γεγονός ότι δεν αναφέρουμε τις γυναίκες που κινδυνεύουν και απειλούνται από ακροτηριασμό των γενετικών τους οργάνων. Δεν αναφέρουμε καθόλου τις γυναίκες, τα κορίτσια που 8-9 ετών τα αναγκάζουν σε γάμο, που είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ένας πλήρης κατάλογος τέτοιων ευάλωτων περιπτώσεων. Αν αφήνω την παράγραφο αυτή να μην είναι για να δηλώσω ότι δεν είμαστε κατά της αρχής, αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει να υπογραμμίζουμε μία μόνο πτυχή του προβλήματος, τότε είμαστε ατελείς. Ίσως θα μπορούσαν να αν συμφωνεί ο εισηγητής και η Επιτροπή μας, να συμπληρώσουμε με μια προφορική τροπολογία την τροπολογία αυτή, ώστε να συμπληρωθούν και οι άλλες περιπτώσεις. Γιατί και αυτές πρέπει να τις υποστηρίξουν. Και αυτήν που αναφέρατε εσείς, σύμφωνοι, αλλά και τις άλλες. Ελπίζω να σας εξήγησα την στάση της ομάδας μου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Στήρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να επιστήσω την προσοχή μας στο ότι με τον κατάλογο αυτό ασφαλών χωρών που αναφέρουμε εδώ, εκτός από την Τουρκία, έχουμε και χώρες της οχι Ιουγκοσλαβίας, χώρες οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι έχουν προχωρήσει περισσότερο, κάποιε λιγότερο. Όλε πάντω έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία προσχώρηση. Και μερικέ φορέ υπάρχουν και θεσμικέ συμφωνίε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτέ. Και υπάρχουν αυτέ οι συμφωνίε γιατί οι χώρε αυτέ ήδη έχουν φτάσει σε κάποιε συγκεκριμένε προδιαγραφέ. Αλλιώ δεν θα είχαν φτάσει να είναι υποψήφιε για προσχώρηση χώρες. Και επειδή πέρασα κι εγώ από αυτή τη διαδικασία, όταν ε, εργαζόμουν στην κρατική υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων, έχει σημασία η προστασία των ευάλωτων ομάδων. Όπως ε, ακούσαμε και πριν, τέτοια προστασία δεν είναι τέλεια πουθενά στον κόσμο. Χωρίς να θέλω να πω με αυτό ότι δεν υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας. Πάντως για τις υποψήφιες αυτές χώρες, αν με τι άλλο, αναμένουμε ότι θα βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση μέχρι να γίνουν μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αναγνωρίζουμε ότι ήδη βρίσκονται σε κάποιο αποδεκτό επίπεδο. Για τελείως δεν θα είχαμε αρχίσει να συζητάμε διαδικασία προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν συμφωνήσαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι χώρες αυτές ανταποκρίνονται σε κάποιες προδιαγραφές, νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό στη συνέχεια να πούμε ότι είναι ασφαλείς χώρες, όπως αναφέρεται στην ε, πρόταση αυτή. Δεν νομίζω ότι βοηθάει το να προσθέτουμε αμφιβολίες εδώ. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για αυτές τις χώρες, να μην είναι καν στη διαδικασία προσχώρησης. Αλλιώς, εφόσον τις κρατάμε στη διαδικασία προσχώρησης, τότε αποδεχόμαστε ότι έχουν φτάσει σε κάποιο καλό επίπεδο και από εκεί και πέρα φυσικά να μένουμε να βελτιωθούν παρετέρω μέχρι την ένταξή τους. Οπότε, συμφωνώ και οι τροπολογίε, ό,τι τροπολογίε έχουμε εδώ, δεν πρέπει με τίποτα να θέτουν υπό αμφισβήτηση το επίπεδο στο οποίο έχουν ήδη φτάσει οι χώρε αυτέ. Ευχαριστώ, δεν βλέπω να ζητάει κανένα άλλο το λόγο. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Κυρία Σάφιν, σωστά. Μπορείτε να μας πείτε από ποιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είσαστε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Home και το τμήμα για το άσυλο πιο συγκεκριμένα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Τα σημειώσαμε. Θα ήθελα να απαντήσω στα κύρια σχόλια που ακούσαμε. Το γεγονός ότι υπάρχει τέτοιος κατάλογος ασφαλών χωρών δεν σημαίνει ότι οι αρχές των χωρών μελών δεν πρέπει ατομικά να εξετάζουν κάθε αίτηση ασύλου. Έπειτα για τις νέες τροπολογίες που σήμερα υποβάλλεται και έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται και η αρχή της ασφαλούς χώρας, η οδηγία προβλέπει ότι σε περίπτωση που υπάρχει σοβαρή πόνια ότι η χώρα δεν είναι ασφαλής για ένα συγκεκριμένο ετούντα, τότε μπορούν να εξεταστούν ειδικέ συνθήκες και προϋποθέσεις. Είδα επίσης ότι μία τροπολογία σας έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ο Ετούν χρησιμοποιεί την ε, ιδέα αυτή το ότι υπάρχει πόνια μια ασφαλούς ε, χώρας και πρέπει να έχει σοβαρές αποδείξεις για το ότι δεν είναι για το συγκεκριμένο ασφαλής ή εν λόγω χώρο. Οπότε δεν έχουμε αλλάξει τίποτα. Οι εγγύσεις έχουν εξεταστεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ιδιαίτερα η απόδειξη για τον ε, σεξουαλικό προσανατολισμό. Φυσικά και πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν οι αρχές ασύλου αποφασίζουν κατά πόσο υπάρχει ή δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο, όπως λέει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. η αποτελεσματική πρόσβαση σε μέτρα διόρθωσης στην περίπτωση που υπάρχει απόρριψη του ασύλου. Η οδηγία λέει ότι δεν υπάρχει αυτόματη τέτοια διαδικασία, αλλά μπορεί να υπάρξει αναστολή είτε μετά από αίτημα του ετούντος ή εξοφίσιο. Τέλος, όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες, σε ένα επεξηγηματικό memorandum η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες που έχουν εντοπιστεί στο memorandum της πρότασης. Οπότε λέμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις ευάλωτες αυτές ομάδες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Σεμπ. Κάποια σημεία ακούστηκαν. Θα ήθελε να σχολιάσει ιδίω για τι μειονότητε, για διάφορε ομάδε που αναφέρθηκαν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Ναι, οπωσδήποτε. Ευχαριστώ του συναδέλφου για τα σχόλιά του. Βλέπω ότι υπάρχει στήριξη για τη συλλογιστική που ακολουθώ στη σύνταξη της έκθεσης ως προς τα συγκεκριμένα εδάφια, γενικώ τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Προφανώς είχαμε πολλές ευκαιρίες να διορθώσουμε τον κατάλογο και θα έχουμε εντός της έκθεσης αλλά η ουσία είναι να υπάρξει στήριξη τη συλλογιστική ε, για το τι λέμε και το πώς θα πρέπει να το κατάλογο κατάλογος ασφαλών χωρών. Δηλαδή, για να έχουμε έναν καταρτισμένο κατάλογο τέτοιων χωρών, θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη μια σειρά από κριτήρια και παράγοντε. και το τι μεταχείριση έχει μια σειρά από ομάδε και μειονότητε. Αυτό μπορεί να συμβαίνει με χώρε που θα βρεθούν ή δεν θα βρεθούν σε αυτόν τον κατάλογο Οπότε υπονοείται ότι το σύστημα θα πρέπει να εξετάζει τις περιπτώσεις ξεχωριστά, αντί να ισχύει συνολικά με μια ομάδα κριτηρίων, προδικάζοντας τις επιμέρους αιτήσει των ε, μεμονωμένων ετούντων. Νομίζω ότι αυτό το ακούσαμε και από τα σχόλια που έγιναν. Τώρα ως προς την προφορική τροπολογία για το να προσθέσουμε κάποιες ομάδες μειονοτικές κατάλογο. Σίγουρα αυτό μπορεί να γίνει, αλλά όπως είπα, η έκθεση δεν έχει τροποποιηθεί για να το λάβει αυτό υπόψη εκ των προτέρων. Σίγουρα πρέπει να το λάβουμε υπόψη στην ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα. αλλά φαίνεται συνολικά ως Επιτροπή να ε, στηρίζουμε την ιδέα του ασφαλούς καταλόγου, του καταλόγου ασφαλών χωρών. Το ζήτημα είναι πώς θα το καταρτήσουμε ως γενικό σύστημα και πώς θα το προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρος, ναι, Έχουμε ακόμα κάποιες διαφωνίες, ε, υπάρχουν κάποιες αποκλήσεις απόψε, αλλά θα ψηφίσουμε έτσι τελειώσουμε μετά το απόγευμα. Να πάμε στο επόμενο σημείο και να σας θυμίσω, συνάδελφοι, ότι στο επόμενο σημείο, 12 παρατέταρτο, έχουμε και προκεκλημένο ε, για την επίσημη ανεπτυξιακή βοήθεια από την ανάλογη επιτροπή του ΩΣΑ. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 8 τα ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστευτες στι τρίτε χώρε. Αυτό συνδέεται με τα προηγούμενα προφανώ. Η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή ΑΦΕΤ και η Υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η δική μας εισηγήτρια, η Μαρίνα Αλμπιόλ, έχει ιδίας γνωμοδότηση ε, έκθεση στην, ε, που θα προσθεθεί στην βασική έκθεση της κυρίας Βερζιά θα ψηφίσουμε για τη δική μας λοιπόν γνωμοδότηση σήμερα το απόγευμα. Καλό θα να τη δείτε. Και τώρα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την Μαρίνα Αλμπιόλ. Μαρίνα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ όλες τις πολιτικές ομάδες και τη Γραμματεία για τη βοηθιά τους. Η αλήθεια είναι ότι παραλάβαμε πολλές τροπολογίες είναι μερικέ οι οποίες βελτιώνουν τη γνωμοδότηση, όπως εκείνες οι οποίες ζητούν την ε, τήρηση του 7 για τις 100 για την ανάπτυξη, άλλες τροπολογίες που αναφέρονται στα παιδιά, στην εκπαίδευσή τους, στην υγεία τους κτλ. Αυτές είναι τροπολογίες οι οποίες, όπως λέω, βελτιώνουν τη γνωμοδότησή μου. Ήθελα να κάνω μια γνωμοδότηση, η οποία δεν θα μείνει στην επιφάνεια, αλλά θα είναι επικριτική για το ζήτημα. Να αναλάβουμε τις ευθύνες που έχουμε και εμείς όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση από τρίτες χώρες. Είναι δύσκολο να φτάσει κανείς σε συμβιβασμό όταν σε 8 παραγράφους οι σοσιαλιστές προτείνουν τη διαγραφή τεσσάρων τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών από τρίτες χώρες όντως παραβιάζονται σε πολλές χώρες, στα κέντρα κράτησης, ότι πολλοί είναι θύματα εκτοπισμού και παράνομων πρακτικών. Δεν ήθελα να φτιάξω μια έκθεση από τα γραφεία απλώς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κλείνοντας τα μάτια στην πραγματικότητα. Εκείνοι όμως δεν θέλουν να αναφερθούμε στην αρνητική δράση των πολυεθνικών, την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε τρίτες χώρες και την εκμετάλλευση ανθρωπίνων και φυσικών πόρων που έχει οδηγήσει σε φτώχεια τόσες πολλές χώρες με αποτέλεσμα να μεταναστεύουν από εκεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Ούτε θέλουν να μιλήσουμε για τα κονδύλια που δίνουμε στην ανάπτυξη για να επηρεάσουμε την οικονομική πολιτική άλλων χωρών, ούτε θέλουν να αναφέρεται η δράση στρατιωτική των χωρών μελών σε τρίτες χώρες που οδηγούν επίσης στη μετανάστευση. Κυρίως βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό ότι θέλουν να διαγραφεί αυτό που αναφέρεται για συμφωνίε μετανάστευση με τρίτε χώρε οι οποίε παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μα αν μη τι άλλο, αυτό είναι το ελάχιστο το οποίο θα έπρεπε να λέει η Επιτροπή μα. Δεδομένη τη κατάσταση, μάλιστα, που βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε και κάνει συμφωνίε με το Μαρόκο και την Τουρκία, όπου οργανώσει όπω η Διεθνή Αμνηστία λέει επανειλημμένα κάθε χρόνο ότι γίνονται φοβερέ παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς, αν μη τι άλλο, θέλουμε να ζητήσουμε να διακοπούν τέτοιες συμφωνίε με χώρες που παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλές λοιπόν τροπολογίες, το μόνο που θέλανε ήταν να αδειάσουν από περιεχόμενο τη γνωμοδότηση αυτή και πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που έχω διαλέξει εγώ ως εισηγήτρια. Οι δύο συμβιβασμοί ελπίζω να προχωρήσουν. Είναι ένας γενικός που μιλάει για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναφέρει τις οικονομικές, πολιτικές και άλλες αιτίε της μετανάστευσης, την προστασία σε ευάλωτες ομάδες ή το θέμα της μετανάστευσης ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στο διάλογο με τρίτες χώρες και υπάρχει και άλλη συμβαστική που αναφέρεται στο χρέος των τρίτων χωρών. Δεν προτείνει την ακύρωση που η ΓΚΟΕ... Αυτό θα ήθελε, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο έτσι βγαίνουν από τη φτώχεια αυτές οι χώρες, προτείνει όμως την αναδιάρθρωση, αν με τι άλλο, του εξωτερικού χρέους. Αυτή λοιπόν είναι η συμβαστική πρόταση δεδομένων των τροπολογιών που μας έφτασαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τους σκιώδεις συζητητές. Πρώτα η κυρία Τερέζα Χιμένες. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Αλμπιόλ για τις εξηγήσεις που μας έδωσε όσον αφορά την ε, έκθεση αυτή και τις τροπολογίες. Στη Λίμπε το Μάρτιο το είχα ήδη πει ότι δεν συμφωνώ με τον ε, τόνο που δίνει στη γνωμοδότηση αυτή η συγγήτρια, συντάκτρια. και την άκουσα και σήμερα που λέει ότι δεν έχει γίνει αυτό, εκείνο, το άλλο. Δηλαδή, τι εννοεί, ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα εδώ, ούτε Λίμπη, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βελτιωθεί η κατάσταση με τους μετανάστες. Νομίζω ότι όλοι έχουμε την ίδια ευαισθησία απέναντι στο θέμα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί όταν λέει ότι από τα γραφεία μας καθόμαστε και κάνουμε εκθέσεις, τέλος πάντων. Εδώ πάντως επικεντρωνόμαστε με την πρόταση αυτή σε πράγματα μη επικοδομητικά κατά τη γνώμη μου. Όλοι είμαστε ευαίσθητοι στο θέμα της μετανάστευσης, τη μεταναστευτική και ανθρωπιστική κρίση. Χτες ήμουνα με το δήμαρχο της Λέσβου, που είναι από τα μέρη όπως και η Λαπεντούσα που έχουν υποφέρει περισσότερο, έχουν πληγεί περισσότερο και πρέπει να λυθεί το πρόβλημα αυτό στη ρίζα του το λένε και εκείνοι. Από εκεί που έρχονται, εκεί πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Γιατί όταν φτάνουν στη Λέσβο, ε, αναγκαστικά περνάνε από μια κόλαση. Για πολλές φορές, πολλοί από αυτούς έχουν χάσει τη ζωή τους. Άρα λοιπόν αυτή η γνωμοδότηση είναι μια ευκαιρία για να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο τίτλος το λέει, ότι μιλάμε για τις χώρες προέλευση. όχι για το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Υπάρχουν άλλε εκθέσει από τη Λίβη και από που αναφέρονται σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Επικεντρωνόμαστε λοιπόν σωστά σε αυτό που γίνεται και εδώ, αλλά σε αυτό που γίνεται και πριν φτάσουν σε εμά. Νομίζω λοιπόν ότι όπως είπα, αντί να μιλάμε για την μετανάστευση φτάνει στην Ευρώπη. Εγώ στην 8 προπολογία ζητάω οι χώρες προέλευσης να βελτιώσουν τα δικαιώματα των ε, μεταναστών και να μπορούν να έχουν θεώρηση πριν φτάσουν σε εμά. Στην τροπολογία 10 λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να λύσουμε το θέμα της λαθροδιακίνησης γιατί πρόκειται για ένα εμπόριο το οποίο αυξάνει τις μεταναστευτικές ροές. Στην παράγραφο 4 επίσης θέλω αλλαγή όσον αφορά τις θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν κάποιες επιχειρήσεις στις χώρες προέλευσης. Και αυτό το συνδυάζω και με την τροπολογία για τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη. Φυσικά και υπάρχουν καταχρήσεις, φυσικά και υπάρχουν πολλά που μπορούμε να καταγγείλουμε, αλλά υπάρχουν και θετικά. Πρέπει να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί απασχόληση και να υπάρξει πλούτος και στις χώρες αυτές. Στην τροπολογία μου 11 ζητάω από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να προωθήσει να δώσει περισσότερη σημασία στην εκπαίδευση για τα παιδιά και εκείνων που έχουν εκτοπιστεί, ζουν σε καταβλισμούς και λέω ότι έτσι εξασφαλίζεται η αξιοπρέπεια και αποκαθιστά το ανθρώπινο δικαίωμα του παιδιού για μια παιδική ηλικία με φροντίδα. Στην τροπολογία 9 πρέπει να υπογραμμίσουμε πώς θα βελτιώσουμε την προσωπική κατάσταση των μεταναστών στους καταβλισμούς, να καταλάβουμε καλύτερα τις προσωπικές τους ανάγκες, ιδιαίτερα των παιδιών των ε, αναπήρων και των γυναικών. Αυτό το θέμα το έχουμε αντιμετωπίσει και εδώ στην προηγούμενη θητεία υπήρχε μια οδηγία για την προστασία των ατόμων αυτών. Ευχαριστώ την εισηγήτρια που έχει συμπεριλάβει πολλές από τις τροπολογίες μας και καταφέραμε να πετύχουμε μια καλή συμβαστική πρόταση που είναι η συμβαστική τροπολογία αριθμός 1. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Περέιρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση που θα ψηφίσουμε το απόγευμα αφορά ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό. Είμαι πεπισμένος ότι με τις ε, συμβαστικές λύσεις που έχουμε βρει και τις τροπολογίες που θα υποβάλλουν ως την ψηφοφορία οι διάφορες πολιτικές ομάδες, η έκθεση αυτή θα είναι μια εύστοχη συνεισφορά της Επιτροπής ΝΤΕΒΕ στην γνωμοδότηση της Καθήλυνα Αρμόδιας Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων. Μετά από τι διάφορε συζητήσει που είχαμε με την εισηγήτρια την κυρία Αλμπιόλ, πιστεύω ότι όλε οι πολιτικέ ομάδε συμμερίζονται τι περισσότερε από τι μεριμνέ τη και αυτό που είδα από την πλευρά των περισσότερων ομάδων, ιδίω των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, την ομάδα SD, είναι επικοδημητικό πνεύμα συνεργασία προκειμένου να υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία όλων των πολιτικών παρατάξεων στην προσέγγιση αυτή του Κοινοβουλίου και με βιώσιμους στόχους. Θέλουμε να ενισχυθεί η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης και θελήσαμε αυτό να αντικατοπτρίζεται και τις μεταναστευτικές μας πολιτικές. Εκεί που δεν συμφωνώ απολύτω με την εισηγήτρια κυρία Αλμπιόλ είναι πω ε, στον τρόπο που αξιολογεί τι τροπολογίε τη ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην όλη διαδικασία. Μάλιστα μου φαίνεται λίγο περίεργο που καταγράφονται εδώ απλώ οι διαφωνίε και αποκλήσει μεταξύ των ομάδων, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια αυτή τη διαδικασία δεν έγινε ούτε μία συνάντηση μεταξύ σκιωδών εισηγητών. Είμαι πεπισμένο ότι μια συνάντηση τέτοιου είδους που ε, έστω και τώρα την έχουμε εδώ στη συνεδρία της Επιτροπής θα είχε συμβάλει να, στο να συνεννοηθούμε καλύτερα και να συμφωνήσουμε σε περισσότερα σημεία. Η γραπτή διαδικασία που προτίμησε να ακολουθήσει η συγκήτρια ε, αναγκαστικά λόγω χρονικών περιορισμών δεν ήταν άνετη. Υποβλήθηκαν προτάσεις το απόγευμα της Παρασκευής, 15 Απριλίου, ε, και οι διάφορες πολιτικές ομάδες είχαν χρόνο να αντιδράσουν ως τη Δευτέρα το απόγευμα. Μεταξύ Παρασκευής απογεύματος και Δευτέρας απογεύματος δεν απολύσει ο χρόνος. Υπάρχουν λοιπόν αποκλήσεις, το διαπιστώνει η συγκήτρια, αλλά πώς μπορεί να μην οργανώνει η συζήτηση των σχεδόν εισηγητών. Και η προθεσμία που διαθέτει στις πολιτικές ομάδες για να αντιδράσουν στις προτάσεις της, Σαββατοκύριακο με μερικές ώρες μόνο, μάλλον μερικές ώρες μόνο με ένα Σαββατοκύριακο στη μέση, δεν αφήνουν ε, χρόνο να τοποθετηθούμε σωστά για ένα θέμα τόσο ευαίσθητο. Θέλω πάντως να ε, καταστήσω σαφές ότι από την πλευρά των σοσιαλιστών και δημοκρατών δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να εντοπίσουμε τις ελλείψεις και τα κενά της ευρωπαϊκής πολιτικής ως προς τη μετανάστευση, τις μεταναστευτικές ροές ή την άφηξη των μεταναστών. Δεν είναι εκεί όμως το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η γνωμοδότηση αυτή έχει ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Η γνωμοδότηση αυτή αφορά τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι το αντικείμενο της έκθεσης. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και αυτό να αναπτύξουμε, όχι άλλα ζητήματα που αφορούν γενικώ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι είναι κάπως καταχρηστικό το κατά πόσον παραμένουμε πιστοί στο αντικείμενο του, της έκθεσης ε, να επηρεάζεται από άλλα σημεία που μπορεί να αφορούν την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Μιλάμε εδώ για τη συνεισφορά της Επιτροπής ΔΕΒΕ που θέλουμε να σεβαστεί τον στόχο της, ε, επιτρο... έκθεσης που θα ετοιμάσει η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, η Επιτροπή ΑΦΕΤ. Και όπως είπα η έκθεση αυτή αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών στις τρίτες χώρες. Πάντως ε, φαίνεται να υπάρχει ε, ε, ικανοποίηση για τις προτάσεις που γίνονται αποδεκτές από την εισηγήτρια, τις προτάσεις της δικές μας. Θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα. Φαίνεται ότι κάποιες πολιτικές ομάδες υπέβαλαν λιγότερες τροπολογίες και ίσως δέχτηκαν και πιο εύκολα για αυτό το λόγο τις δικές της συμβαστικές τροπολογίες. Οι δικές μας όμως προτάσεις ήταν αυτές και ελπίζω ότι παρά τον όγκο των τροπολογιών θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια καλύτερη γνωμοδότηση τελικά με τις αλλαγές που έχουμε προτείνει. Και τώρα η εισηγήτρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα από την Καθήλυνα μου Επιτροπή, κυρία Βεζιά. Αλλά θα σας δώσω τον λόγο θα ακούσουμε και τους υπολοιπούς συμμιλητές αν δεν σα πειράζει. Ο κύριος Γκέρενς. Θέλετε το λόγο τώρα, κύριε Βερζιά. Επειδή μόλις στάσατε, ήθελα να περιμένω να δω μήπως θέλετε να ακούσετε πρώτα τους συναδέλφους. Αλλά θέλετε να πάρετε το λόγο αμέσω, προφανώς έχετε κάπου να πάτε κιόλα, κυρία Βερζιά. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα. Σήμερα το πρωί εξέτασα τις τροπολογίες και είδα πώς θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιες συμβαστικέ. Ε, λύσεις και είμαι και μέλο στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που συζητάμε τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματο Ασύλου. Τα θύματα αυτά είναι αλληλένδετα, όπω ξέρετε. Οπότε, μόλι άκουσα την ε, εισήγηση του σοσιαλιστή συναδέλφου, αλλά όπω ξέρετε, κυρία Αλμπιόλ, ήταν παρούσα σήμερα στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ξέρω λοιπόν πώ έχει προχωρήσει το θέμα. Και επίση πρέπει να πω ότι έχω δει τι τροπολογίε σα και τι συμβαστικέ λύσει που έχουν ποταθεί Θα ήθελα λοιπόν να επιμείνω σε κάποια σημεία. Για μένα ένα μέγιστο πρόβλημα είναι το πώς θα συντάξουμε την έκθεση αυτή. Δεν θέλουμε να είναι η επανάληψη τη έκθεση που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα και που αφορά ακριβώ τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Έχουμε να κάνουμε με μια έκθεση τη Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία θα ψηφιστεί στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και που αφορά ακριβώ τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη θέση των μεταναστών σε τρίτε χώρε. Οι προβληματισμοί μας λοιπόν είναι να ξαναδούμε το θέμα της μετανάστευσης σε ένα τοπίο διεθνές δεν θέλουμε απλώς να συγκεντρωθούμε στην οπτική γωνία των Ευρωπαίων, αλλά να δούμε συνολικά την εικόνα των μεταναστευτικών πολιτικών στο σύνολό τους. Αυτό είναι το αντικείμενο της έκθεσης που υπέβαλα. Θέλουμε να δούμε πώς το ζήτημα της, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών ιδιαίτερως ε, διαμορφώνεται σε τρίτες χώρες και πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές εντάσσονται στις διεθνείς πολιτικές γενικότερα και στις αναπτυξιακές πολιτικές και μπορούν να βοηθήσουν να βελτιωθεί η θέση των μεταναστών και η γενικότερη κατάσταση. Στην Επιτροπή Ντροά έχουμε περίπου 300 τροπολογίες να εξετάσουμε. Από μόνη της αυτή είναι μια μικρή πρόκληση. Όμω η συζήτηση που είχαμε το πρωί ήταν, ε, πιστεύω, ιδιαίτερη, ε, ιδιαίτερα επικοδομητική Ενώ όλοι του Έχουμε την ίδια επιθυμία να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συνένεση, όσο το δυνατόν ευρύτερη. Πραγματικά χαίρομαι που η Επιτροπή Ανάπτυξη, η Επιτροπή σα, θα εγκρίνει εν ευθέτω χρόνο αυτέ τι τροπολογίε, ελπίζω, δηλαδή μετά τη λήξη τη ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών συμβιβασμού και έτσι θα προλάβουμε να εντάξουμε τι τροπολογίε τη Επιτροπή ΔΕΒΕ στι δικέ μα συμβαστικέ τροπολογίε. Συμμεριζόμαστε, πιστεύω, κάποιε ε, από τι ανησυχίε μα που είναι κοινέ. Οπότε μου φαίνεται καθοριστική σημασία το εξή. Εάν οι πολιτικές μάλλον οι πολιτικές αναπτυξιακές βοήθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιούνται επαρκώς και να ξαναδούμε ακριβώς την αναπτυξιακή μας βοήθεια. Υπάρχει μια ε, πρόκληση για την οποία πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη εγρήγορση. Αυτή είναι περίπου η δική μου η προοπτική στα πράγματα και είμαι τελείως ανοιχτή. Είμαι τελείως πρόθυμη να συνεργαστούμε διότι τα θέματα αυτά είναι αλληλένδετα και οι αναπτυξιακές πολιτικές είναι καθοριστική σημασία για τα θέματα αυτά, αλλά μην ξεχνάμε ότι στην έκθεση αυτή επικεντρωνόμαστε σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. το πρόβλημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών. Μην ξεχνάμε ότι σε πολλέ από τι χώρε που τι αφορά η αναπτυξιακή μα πολιτική υπάρχουν ελάχιστε ε, από αυτέ που έχουν συγκεκριμένε πολιτικέ για τα δικαιώματα των μεταναστών. Δεν λαμβάνουν καν υπόψη του αυτή τη μέρημνα. Μιλάω για τη Σύμβαση τη Γενέβης και το σεβασμό του δικαιώματος ε, αίτηση ασύλου. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο θέλουμε να προσεπιστούμε και θέλουμε να επιμένουμε σε αυτό. Νομίζω ότι γενικώ υπάρχει συνένεση γι' αυτό έτσι κι αλλιώ στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Συμφωνούμε ότι ζητάμε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να έχει μια συνολική λύση. Οπότε προφανώ και πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ διαφορετικών κοινοβουλευτικών επιτροπών, γιατί δεν μπορεί κάθε επιτροπή να προτείνει μια διαφορετική πολιτική. Ωραία. Σαρ Βιόρεντς, ο επόμενο Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την κυρία Βερζιά που παρουσίασε τι απόψει της. Αυτό που με απασχολεί εμένα πρώτα απ' όλα είναι η θέση και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι συμφωνούμε στην Επιτροπή μας ότι θέλουμε να υπάρχει ανθρώπινη αντιμετώπιση με αξιοπρέπεια των ε, μεταναστών βάσει των συμφωνιών που έχουμε συνυπογράψει και των συμβάσεων. Βέβαια, ο λόγος των πολιτικών μας ρίχνει λάθη στη φωτιά πολλές φορές, αντί να κάνουν το αντίθετο. Κάτι που είναι απαράδεκτο. Και αυτό ακριβώ είναι το οποίο δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τη δικιά μα τη δουλειά. Δεύτερον, με μια γνωμοδότηση προ μια άλλη επιτροπή που είναι αρμόδια επί τη ουσία, εννοείται ότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε όλα τα στοιχεία που σκεφτόμαστε για να λυθούν οι κρίσει που αναφέρονται στην έκθεση. Όμω θέλω να αναφερθώ στην παράγραφο 8 που τροποποιήθηκε με συμβαστική, αν δεν κάνω λάθος. Και έχει να κάνει με την ακύρωση του εξωτερικού χρέους. Σίγουρα το χρέος βαραίνει πάρα πολύ, αποτελεί υποθήκη για την ανάπτυξη των χωρών. Αλλά για να υπάρχει χρέος σημαίνει ότι κάποιος δανείζει. Κάθε φορά που κάποιος δανείζεται, κάποιος τον δανείζει. Αυτό που με ενοχλεί λοιπόν εμένα στην παράγραφο αυτή 8 και στη συμβαστική είναι ότι δεν αναφέρεται καθόλου η ευθύνη αυτού που δανείζει έτσι με ευκολία. Έχει και αυτός ευθύνη, διότι ακριβώς ανεβάζει το παθητικό της χώρας την οποία δανείζει, άρα ενισχύει αυτή την υποθήκη που αναγκαστικά βάζει χώρα. Οπότε ναι, εξωτερικό χρέος ακύρωση ναι, αλλά εφόσον υπάρχει μια νέα προσέγγιση. Και εξηγούμε. Αντί να λέμε απλώ και μόνο ακύρωση του εξωτερικού χρέου, οι χώρες πιστωτέ και τα διεθνή, οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να πούνε ναι, συμφωνούμε να παραιτηθούμε από τα χρήματα που δανείσαμε στη χώρα Χ. Υπό τον όρο ότι το χρέος αυτό που δεν θα πληρωθεί στον πιστωτή θα αλλάξει και θα γίνει χρέος που θα αποπληρωθεί σε τοπικό νόμισμα. Δηλαδή δεν θα επιστρέφεται στον πιστωτή, αλλά θα προσφέρεται για την βελτίωση των υποδομών στην λόγω χώρα, εκπαίδευση, υγεία, πρόσβαση στο νερό κλπ. Σε αυτή την περίπτωση βάζουμε το κράτος μπροστά στις ευθύνες του. Δεν διαγράφουμε απλώς και πλήρως το χρέος, αλλά κάνουμε αυτό που λέει και η τροπολογία, ότι κάνουμε δηλαδή κάτι πολύ συγκεκριμένο προς όφελος της χώρας. Και βάζουμε μπροστά στις ευθύνες της για να αναλάβει την ανάπτυξή της η ίδια η χώρα. Αν τώρα η Επιτροπή, γιατί δεν ξέρω ακόμα για την ψηφοφορία για το απόγευμα. Αν συμφωνούμε να αντιμετωπίσουμε έτσι το θέμα και δέχεστε να κάνουμε μια δική έκθεση για το χρέος που μπορεί να μετατραπεί σε αναπτυξιακή βοήθεια, τότε ευχαρίστως να προτείνω να ψηφίσει η ομάδα μου υπέρ της συμβαστικής που περιλαμβάνει το σημείο αυτό 8. Ευχαριστώ πολύ κυρία Θαουτάλα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω και εγώ ότι ακούσαμε πολύ καλές ε, συμβουλές από τους συναδέρφους ε, Περέιρα και Βερσιά. Να εμείνουμε δηλαδή στον τίτλο δηλαδή που έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την μετανάστευση. Είναι ένα θέμα που συνδέεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και συμφωνώ ότι δεν πρέπει να το συνδέσουμε με ε, άλλα θέματα. Θα πρέπει να φροντίσουμε να συμπεριλαμβάνονται όλα τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εδώ. Αναφερόμαστε στις ανάγκες περιθωριοποιημένων ομάδων. Γίνεται αναφορά στην αντιμετώπιση των αιτιών της μετανάστευσης. Έχω όμως και μία ερώτηση σχετικά με ε, την συμβαστική τροπολογία 8. Νομίζω ότι η πρώτη πρόταση είναι υπερβολικά επιτακτική που αναφέρεται στην διαγραφή του χρέους των χωρών αυτών και άλλων αναπτυσσόμενων χωρών τα υπόλοιπα μπορεί να είναι σωστά και μπορεί να υπάρξουν κάποιες καινοτόμες λύσεις όπως αναφέρθηκε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολύ κομψή η διατύπωση της σύμβαστικής αυτής τροπολογίας. Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. Πάντως, ε, σίγουρα οι ε, συμβιβαστικές τροπολογίες έχουν βελτιώσει την ποιότητα αυτής της ε, γνωμοδότησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να τονίσω κάποιες ιδέες που θα ήθελα να καλέσω ε, την εισηγήτρια να συμπεριλάβει στις ε, συμβαστικές ε, τροπολογίες. Η αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεχίσει να έχει ως βασικό στόχο την εκρίζωση της φτώχειας. Δεύτερον, θεωρώ ότι η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις αιτίε της μετανάστευσης σε πολιτικούς, οικονομικούς και ε, περιβαλλοντικούς λόγους. Και θα ήθελα να τονίσω ότι τα προγράμματα ε, αναπτυξιακής βοήθειας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για στόχους ελέγχου της μετανάστευσης ε, και διαχείρισης των συνόρων. Τέλος, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την σχέση ανάμεσα ε, στην αναπτυξιακή βοήθεια και τη μετανάστευση χωρίς να αρνούμαστε ότι η ε, αναπτυξιακή βοήθεια μπορεί να μετριάσει τις ε, συνέπειες της αναγκαστικής μετανάστευσης βοηθώντας την επίλυση διαφορών και προωθώντας το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάνω την εισηγήτρια να συμπεριλάβει όλες αυτές τις ιδέες. Σας ευχαριστώ πολύ και να κάνω κι εγώ μια παρατήρηση σχετικά με την παράγραφο 8. Μάλλον ε, δεν θεωρώ ότι οι καταχρήσεις ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων ε, θα σταματήσουν λόγω της βοήθειας, της οικονομικής μας βοήθειας προς κάποια καθεστώτα. Δεν θα πρέπει πάντα να θεωρούμε ότι συνδέονται αυτά και θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να επικρίνουμε ε, τα καθεστώτα όταν ε, αυτό είναι σωστό. Γνωρίζουμε ότι επίσης ε, δεν δαπανούν όλες οι χώρες τα χρήματα που τους δίνονται για οργανώσεις πολιτών, συστήματα υγείας και την εκπαίδευση. Είδαμε τι έγινε στον Παναμά. Είδαμε δηλαδή τι γίνεται όταν διάφοροι άνθρωποι προσπαθούν να αποσύρουν τα χρήματά τους ε, από τον δημόσιο έλεγχο. Έχουμε εδώ εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Νομίζω δεν θέλει να πάρει το λόγο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Αλπιδόλ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για αυτά που είπατε και για την επικοδομητική σας στάση. Λοιπόν, ποια είναι τα σχόλιά μου. Για όλους μας είναι ξεκάθαρο ότι μέσα σε μια γνωμοδότηση δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε το θέμα της μετανάστευσης. Πρέπει να περιοριστούμε στα ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστευση τρίτες χώρες. Αυτό είναι ο τίτλος, όντως. Για όλους μας είναι ξεκάθαρο. Η διαφορά μας όμως έγινε μέσα σε αυτή τη γνωμοδότηση με αυτό τον τίτλο κατά πόσο έχει θέση ή όχι κριτική απέναντι στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέναντι σε τρίτες χώρες. Εδώ είναι που διαφωνούμε. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δούμε μέσα αυτή τη γνωμοδότηση πώς η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των πολυεθνικών, οι στρατιωτικές παρεμβάσεις, πώς όλα αυτά επηρεάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μετανάστευση σε τρίτε χώρες. Μετά τη συζήτηση λοιπόν που είχαμε εδώ είναι ξεκάθαρο ότι παρόλο που ξεκινήσαμε από αρκετά διαφορετικές θέσεις, καταφέραμε να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές θέσεις και έτσι να προχωρήσει η γνωμοδότηση αυτή. Οπότε, σας ευχαριστώ όλους. Για το θέμα του χρέους τώρα. Πάνω σε αυτό μίλησαν οι περισσότεροι. Ευχαριστώ τον κύριο Γκέρενς. Σωστό αυτό που λέει. Όντως, είναι ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή μας ή να εκπονήσουμε έκθεση για το θέμα της ε, ακύρωσης του χρέους, γιατί είναι κάτι που όλους μας ενδιαφέρει. Αλλά όσον αφορά την γνωμοδότηση, δεν ξέρω τι περιθώριο έχουμε. Και αν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε μια προφορική τροπολογία ή να τροποποιήσουμε λίγο τον, ε, τη συμβαστική πρόταση που περιλαμβάνει αυτή την παράγραφο, ώστε να συμπεριλάβουμε το πνεύμα του κύριου Γκέρενς, δηλαδή ότι με την ακύρωση του χρέους μπορούμε τα χρήματα αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε για ανάπτυξη. Τίποτα άλλο και σας ευχαριστώ πολύ όλους. Θα ψηφίσουμε γνωστό θέμα αυτό. Α, κυρία Βερσιά, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εάν όχι, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ε, από ό,τι κατάλαβα υπάρχουν πολλές τροπολογίες για την έκθεσή σας. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ σημαντική. Επίσης βλέπω ότι σήμερα έχετε οργανώσει ε, συνέντευξη τύπου με διάφορους ε, συναδέρφους ε, σχετικά με την σεξουαλική βία στο Τσάντ. Και νομίζω ότι θα ενδιαφέρει τους ε, συναδέρφους να ακούσουν περισσότερα για το θέμα αυτό. Μιλήσαμε για ε, θέματα φίλου σήμερα. Ε, πάντως χαιρόμαστε για τη συνεργασία μαζί σας και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σας εύχομαι καλή επιτυχία κατά τη συνέντευξη τύπου. Ευχαριστώ πολύ. Θα προχωρήσουμε τώρα στο σημείο νέα της ημερησίας διάταξης. Έχουμε μια προσκεκλημένη. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Ελπίζω λοιπόν ότι θα παραμείνουν ε, στην αίθουσα οι συνάδελφοι. Πρόκειται για το σημείο 9 της ημεσίας διάταξης ε, και υπάρχει έγγραφο στους φακέλους σας στο σημείο 9 ε, θα βρείτε ένα έγγραφο του Γερμανικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης στο σημείο 9 λοιπόν, αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Κίνησης Αντίληψης για την Ανάπτυξη. Συνάδελφοι, όπως είπα, αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα για την Επιτροπή μας. Κατά την τελευταία συνάντηση ενημερώσαμε τους συναδέρφους ότι υπό το φως των στόχων ε, βιώσιμης ανάπτυξης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θέλει να αναθεωρήσει την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη. Ε, πολλοί συνάδελφοι δεν ε, βρίσκονταν στο Κοινοβούλιο όταν υπεγράφει η κοινή αντίληψη το Δεκέμβριο του 2005. Υπεγράφει από τους Προέδρους ε, Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής και, και αργότερα και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Και ήταν το πρώτο έγγραφο που θέσπιζε μια ενιαία σειρά αρχών σχετικά με το πώς θα πρέπει να λειτουργεί η πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και γενικά από το 2005 λοιπόν ε, έγινε σημαντική προσπάθεια να υπάρξουν κοινέ δράσει και κοινό προγραμματισμό σε διάφορε χώρε ώστε η αναπτυξιακή βοήθεια να έχει το μέγιστο δυνατό αντίκτυπο. Ε, έχουν περάσει όμως πάνω από 10 χρόνια από το 2005 και Ήμασταν πολύ φιλόδοξοι τότε, είχαμε την ε, εκστατεία για την εκρίζωση της στόχιας, ε, είχαμε διάσκεψη κορυφής ε, όπου όλοι υποσχέθηκαν ότι θα δίνουν το 0,7% του προπολογισμού τους σε συναρτησιακή βοήθεια. Τώρα, τόσα χρόνια μετά, είχαμε την οικονομική κρίση, έχουμε περισσότερες συγκρούσεις, περισσότερη αστάθεια και πιο απεσιόδοξη οπτική του κόσμου σήμερα από ό,τι είχαμε το 2005. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα αναθεωρήσει την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη, θα ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση από τον Μάιο μέχρι τα τέλη Αυγούστου και Κατόπιν θα παρουσιάσω στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο μια νέα πρόταση για την κοινή αντίληψη. Σήμερα το πρωί οι συντονιστέ συμφώνησαν η Επιτροπή μα μέσα στου επόμενου μήνε να συντάξει έκθεση για να επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να συμβάλλει στην ε, αναθεώρηση τη Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη. Ε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό ε, και θα ε, διαμορφώσει το σύνολο της ε, πολιτικής ε, ανθρωπιστικής βοήθειας. Χαίρομαι που έχουμε εδώ σήμερα την κυρία Κριστίν Χακενές από το Γερμανικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης. Είναι πρωτοπόρο το Ινστιτούτο, διότι πριν από οποιονδήποτε άλλο εκπώνησαν έγγραφο σχετικά με το ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει η κοινή αντίληψη. Γι' αυτό θα ρωτήσω το λόγο για να μας εξηγήσει. Παρακαλώ, Κριστίν. Um, Γεια σας. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε για αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση και που μου επιτρέψατε να πάρω μέρο στην όλη αυτή ε, διαδικασία διαβουλεύσεων σε τόσο έγκαιρη φάση των διαπραγματεύσεων. Η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης μόλις τώρα αρχίζει. Πιστεύω ότι θα είναι μια σημαντικότατη συζήτηση για την αναπτυξιακή πολιτική, διότι η αναθεωρημένη κοινή αντίληψη προφανώ θα καθοδηγήσει τι αναπτυξιακέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα ένα-δύο χρόνια. Για τα επόμενα μάλλον χρόνια. Βρισκόμαστε σε μια φάση μεταβατική. Εσωτερικώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια σειρά από φαινόμενα κρίση που πρέπει να αντιμετωπιστούν μαζί. Η οικονομική, ε, στα κράτη-μέλη λόγω χάρη και ο λαϊκισμός ή η κρίση των προσφύγων. Αυτά δεν είναι μόνο εσωτερικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται να έχουν αντίκτυπο στο πώς γίνεται αντιληπτή η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις χώρες εταίρους. Και επίσης επηρεάζουν και την αξιοπιστία αλλά και το θεμητό της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής. Ταυτόχρονα μαζί με αυτές τις εγχώριες συζητήσεις που γίνονται έχουμε να αντιμετωπίσουμε και κάποιες προκλήσεις στο διεθνές προσκήνιο που και αυτό μεταβάλλεται. Οι κλιματικές αλλαγές, η ε, υποβάθμιση της βιοπικιλότητας, οι αλλαγές και η αύξηση του ποσοστού ένδυας στις αναψώμενες χώρες, ο περιορισμός του πολιτικού περιθωρίου σε κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες και η αυξανόμενη αυστάθεια και το ευάλωτο της κατάστασης όχι μόνο στην άμεση ευρωπαϊκή γειτονιά αλλά και ακόμη πιο μακριά. Σε αυτό λοιπόν το γενικό τό των εσωτερικών προκλήσεων και των εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις ερχόμενες εβδομάδες και μήνες θα συζητήσουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις υπηρεσίες εξωτερικής δράσης των κρατών μελών το ρόλο της αναπτυξιακής πολιτικής στο ευρύτερο ε, πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να βασιστούμε στη συζήτηση αυτή στα εξή θέματα. Τι μπορούμε να κάνουμε με την αναπτυξιακή πολιτική και πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις κρίσεις αλλά και να συμβάλλουμε στην ε, βιώσιμη αναπτύξη παγκοσμίω. Και πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία των διαφορών τομέων αναπτυξιακής πολιτικής μας για να υπάρχει βιωσιμότητα σε όλου τους τομείς με εμπόριο, ανθρωπιστική βοήθεια ή την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Νομίζω ότι ο προγραμματισμός της αυτή στη φάση αυτή που είναι τόσο ε, έγκαιρη είναι πολύ καλό για να δείξουμε και στου Ευρωπαίου πολίτε αλλά και στου ε, εξωτερικού μα εταίρου ότι παρά τι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εντό Ευρωπαϊκή Ένωση η αναπτυξιακή μα πολιτική ε, με μεγάλη σοβαρότητα μπορεί να επιτρέψει συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων φορέων. Ένα πρώτο ζήτημα λοιπόν είναι και ήταν η κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως υπογράφηκε το 2005-2006 και τι έχει πετύχει. Για πρώτη φορά τότε θέσπισε κοινού στόχου και κατευθυντήριε γραμμέ για την αναπτυξιακή πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Με, όλα τα αρμόδια, με όλου του αρμόδιου φορεί των κρατών μελών αυτό. άφησε την προβολή τη αναπτυξιακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αποστείλει το μήνυμα ότι η αναπτυξιακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι παραπάνω από το σύνολο του τι κάνουν τα κρατημέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Έχει επηρεάσει τι όλε διαβουλεύσει για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και κυρίω για τα όργανα αναπτυξιακή βοήθεια γύρω στο 2007. Επίση έχει καθορίσει και διαμορφώσει τι αναπτυξιακέ πολιτικέ των κρατών μελών και έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση τη επίδραση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο διεθνέ προσκήνιο. Επίσης είναι σαφές ότι τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, το έγγραφο είναι του 2005, τα τελευταία ένα-δύο χρόνια λοιπόν, δεν είναι πια τόσο επίκαιρη η πολιτική όπως είχε διαμορφωθεί παλιότερα. Στα πλαίσια τη κοινή αντίληψη συζητιέται ποια είναι η πολιτική των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και της Ευρωπαϊκή Επιτροπής και έχει αντικατασταθεί από την Agenda for Change όπως ονομάστηκε, το θεματολόγιο για την αλλαγή. Εδώ ε, αυτό συνδυάστηκε με τις συζητήσεις για τους στόχους της χιλιετίας και σαφώς υπάρχει ανάγκη για κάποιες θεμελιώδεις ε, αλλαγές και αναθεωρήσεις. Η νέα κοινή αντίληψη θα πρέπει και πάλι να είναι μια ισχυρή πολιτική δήλωση με γενικέ κατευθύνσει και μια στρατηγική θεώρηση για την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική. Θα πρέπει να είναι ένα σύντομο έγγραφο που να καταγράφει απλώ τι προτεραιότητε και τι βασικέ αρχέ τη ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική, αλλά να μην περνάει σε ιδιαίτερε λεπτομέρειε. Θα χρησιμοποιήσω το επόμενο πεντάλεπτο ή εξάλεπτο που έχω για να δείξω κάποια ζητήματα που αφορούν εμένα και του συναδέλφου μου από το Γερμανικό Ινστιτούτο για την και Πολιτική και τα οποία πιστεύω θα μπορούσαν να έχουν ε, ένα σημαντικό ρόλο στην όλη συζήτηση. Πρώτον, είναι ε, σαφέ ότι το θεματολόγιο για την ανάπτυξη που συμφωνήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, το διάστημα 2020-2030, θα μπορούσε να είναι ένα πλαίσιο για, τον, ε, για την έκοινη αντίληψη ατζέντα τη αλλαγή, το θεματολόγιο τη αλλαγή. Θα μπορούσε να καθορίσει προτεραιότητε για τι θεσμικέ αναπτυξιακέ πολιτικέ και το τι κάνουν δημοκρατικέ ε, κυβερνήσει για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Αυτό είναι πολύ καλό σημείο αφετηρία για την όλη συζήτηση, αλλά στο πλαίσιο τη ατζέντα 2020-2030 και με του στόχου που συμφωνήθηκαν για τι κλιματικέ αλλαγέ στο Παρίσι το περασμένο φθινόπωρο, θα ε, είναι σαφέ ότι η νέα κοινή αντίληψη θα πρώτα λάβει και αυτά υπόψη. Επίση, πρέπει να διαμπρίνουμε του στόχου τη Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Πολιτική και να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στι διεθνεί προκλήσει, το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει στην ενισχυμένη συνεργασία με τι πλουσιότερε και αναπτυγμένε χώρε, ιδίω τι χώρε μέσου εισοδήματο, διότι οι χώρε αυτέ είναι πλέον 104 και είναι υπεύθυνο για το 30% του διεθνούς ΑΕΠ. Όμως, στο έδαφο του βρίσκεται και ο μισό πληθυσμό φτωχών ανθρώπων, πολιτών του κόσμου. Και επίση είναι υπεύθυνε για εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Μιλάμε για χώρε ε, πολύ διαφορετικέ μεταξύ του, πολύ διαφορετικέ κατηγορίε και ομάδε, αλλά είναι και πολύ ενδιαφέροντε εταίροι για να αντιμετωπίσουμε διεθνεί προκλήσει και να έχουμε συνεργασία μαζί τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αλλάξει τις πολιτικές της για τις σχέσεις της με τις χώρες μεσοσοδήματος και το θεματολόγιο της αλλαγής έχει ε, προβλέψει την αρχή της διαφοροποίησης, της διαφοροποιημένης προσέγγισης. Στα πλαίσια του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου επίσης, η βοήθεια στις χώρες ανώτερου μέσου έχει μειωθεί η περικοπή. Και ταυτόχρονα, ε, μέσα με τις συζητήσεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνονται σχετικές συζητήσεις σε πολλά κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή επανακαθορίζουν τι δράσει του και τη συνεργασία του με τι χώρε μέσω εισοδήματο. Οι συζητήσει λοιπόν για την κοινή αντίληψη είναι ακριβώ επίκαιρε και σκόπιμε, διότι μπορούν να επιτρέψουν να θέσουμε τα θεμέλια για μια συνένεση μεταξύ θεσμικών οργάνων και κρατών μελών για το πώ πραγματικά να προχωρήσουμε τι σχέσει μα με τι χώρε αυτέ και να, ε, καθορίσουμε, να χαράξουμε συγκεκριμένε στρατηγικέ για τη συνεργασία μα. Οι συζητήσει για τη συνεργασία με τι χώρε μέσω εισοδήματο ήταν κάπω σε αμυντική στάση τώρα, διότι ασχολούνταν περισσότερο με το πώ, πότε και πόσο να περικόψουμε την αναπτυξιακή βοήθεια. Ενώ το βασικό ερώτημα που έπρεπε να θέσουμε είναι πώ να συνεργαστούμε με τι χώρε αυτέ για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη διεθνώ και το κατά πόσο η αναπτυξιακή βοήθεια είναι ένα βασικό στοιχείο τη συνεργασία με τι χώρε αυτέ. Θα πρέπει λοιπόν να καθορίσει ένα τεξιακό πακέτο που να συμπεριλαμβάνει το εμπόριο, το κλίμα και άλλου στόχου και να είναι ελκυστικό για τι χώρε αυτέ ώστε να προχωρήσουν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα, το θεματολόγιο 2020-2030 είναι επίση ένα σημαντικό σημείο αναφορά για τη συνεργασία μα με τι χώρε αυτέ και εάν η Ευρώπη πραγματικά υλοποιεί σωστά το θεματολόγιο αυτό με σοβαρότητα και συνέπεια στι εξωτερικέ τη πολιτικέ, τότε οι χώρε αυτέ θα είναι καθοριστικοί μα εταίροι σε αυτή τη συνεργασία. Το τρίτο μου σημείο έχει να κάνει με την ε, συνεργασία μας με τα πιο ευάλωτα κράτη, αυτά που επηρεάζουν πάρα πολύ και τον όλη συζήτηση για την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη, διότι η ασφάλεια και το ευάλωτο είναι πολύ πιο σημαντικά και κρίσιμα θέματα από ό,τι ήταν το 2005 και 2006 όταν το θέμα πρώτο συζητήθηκε. Οι προβλέψει είναι ότι στο 2030 ο μισό πληθυσμό του κόσμου που βρίσκεται σε κατάσταση ένδυα θα επηρεάζει την διαμόρφωση και την πολιτική των ευάλωτων κρατών. Πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον μπορούμε αυτή την αδυναμία των κρατών να την αντιμετωπίσουμε, να προβλέψουμε διενέξει και να του παράσχουμε μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Αυτό θα είναι κάτι που θα επηρεάσει η πολιτική μα αντίληψη και τι σχετικέ συζητήσει. Πρέπει να δούμε πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα προάγει μόνο στόχου βραχυπρόθεσμου για την ασφάλεια και τη σταθερότητα, αλλά και μακροπρόθεσμα με την τη βοήθεια, στερίζοντα του δημοκρατικού θεσμού. Φαίνεται λοιπόν να υπάρχει μια <coughs> τάση να χρησιμοποιείται η αυτοεξήγηση βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να προάγει του βραχυπρόθεσμο στόχου ασφάλεια και σταθερότητα. Όμω, υπό το φω τη επιδείνωση τη κατάσταση ασφάλεια σε έναν μεγάλο αριθμό χωρών, όχι μόνο στην άμεση γειτονιά μα, φαίνεται ότι αυτό είναι σημαντικό και μα απασχολεί μακροπρόθεσμα το τι θα γίνει. Οι μεταρρυθμίσει του τομέα ασφάλεια, λοιπόν, θα πρέπει να συμβαδίσουν με τη στήριξη των δημοκρατικών θεσμών και τη δημοκρατική διακυβέρνηση, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει μακροπρόθεσμα την σταθερότητα και όχι μόνο βραχυπρόθεσμα. Το άλλο μεγάλο θέμα, σε σχέση με τη συνεργασία μας και τα ευάλωτα κράτη, θα επικεντρωθεί στη σχέση μεταξύ αναπτυξιακής βοήθειας και ανθρωπιστικής. Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη αφορά και την ε, ανθρωπιστική βοήθεια, όπως και καταρτιστεί το 2008. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη πρέπει να καθορίσει μια σχέση και με την ανθρωπιστική βοήθεια. Και είναι ε, απαραίτητο αυτό. Τελευταίο και τέταρτο σημείο συζητήσεις για την ε, συνοχή της πολιτικής μας. Αυτό θα είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης. Η πολιτική, η κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη θα πρέπει να βασίζεται σε μια ευρεία συνένεση που να είναι προτεραιότητα στην ε, ευρωπαϊκή ατζέντα. Ένα από τα βασικά διδάγματα όμως των συζητήσεων ως τώρα για την ασφάλεια και την ε, ανάπτυξη έχουν να κάνουν με το ότι η αναπτυξιακή πολιτική δεν μπορεί να κάνει πολλά για τη συνοχή των πολιτικών εάν οι υπόλοιποι πολιτικοί τομείς δεν δείχνουν διάθεση να συνεργαστούν με τον αναπτυξιακό. Πριν από μία εβδομάδα, την Τετάρτη νομίζω τη περασμένη εβδομάδα, συζητήσαμε με την είπατε εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Φεντερίκα Μογερίνη, για την Ευρωπαϊκή Στατηγική Εξωτερικών Σχέσεων και Ασφάλειας. Στην ομιλία της η κυρία Μογερίνη στεναρά υπερασπίστηκε την ιδέα ότι η νέα μας κοινή αντίληψη θα πρέπει να είναι μια διεθνής στρατηγική, όχι μόνο για τις εξωτερικές σχέσεις και την ασφάλεια, αλλά και για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρύτερα, μαζί και σε αυτά και η αναπτυξική μας ε, βοήθεια και πολιτική. Έτσι λοιπόν φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιστεύει σταθερά ότι συνολικά η αναπτυξική βοήθεια διεθνώ γίνεται μια σημαντική παράμετρο τη ευρωπαϊκή πολιτική εξωτερικών σχέσεων και θα επηρεάσει την διεθνή μα στρατηγική. Αυτό ε, θα καθορίσει και τα ζητήματα συνοχή. Εάν το θέσουμε διαφορετικά δηλαδή, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να προωθήσουμε την πολιτική σύνοχη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, εάν αυτή είχε ενταχθεί συνολικά στη στατική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, έτσι είχε καθοριστεί και η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη. Και τρεις-τέσσερις παρατηρήσεις για να ολοκληρώσω. Όπως είπα αρχικά, η συζήτηση για την κοινή αντίληψη θα είναι καθοριστική σημασία, διότι θα, θα διαμορφώσει το μέλλον τη εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω στην αναπτυξική τη πολιτική για τα ερχόμενα χρόνια. Και θα επηρεάσει τι συζητήσει για τι μεταρρυθμίσει των εργαλείων χρηματοδότηση στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020. Είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσουμε τη σωστή κατεύθυνση και στο μέλλον των ευρωπαϊκών σχέσεων με τι χώρε τη Αφρική, τη Καραϊβική και του Ειρηνικού. Και αυτά ε, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φάση διαπραγματεύσεων και είναι σημαντικό πώ θα οργανωθεί όλη η διαδικασία. Δηλαδή, πέραν των ε, συνηθισμένων διαδικασιών, είναι σημαντικό να αναλάβουμε δράση και να προσκαλέσουμε εταίρους από την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Ασία να μα αναπτύξουν τι απόψει του και να μα πούν τι περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Αναπτυξία και Πολιτική και πώ θα ήθελαν να αισθανθούν με την Ευρωπαϊκή Πολιτική τη ανάπτυξη για να δουν και να μας πούν πώ θα του χρησιμεύσει στο μέλλον. Στο Γερμανικό Ινστιτούτο Ανάπτυξη. και με τους εταίρους μας, ανυπομονούμε για τις όλες τις συζητήσεις και πραγματικά δεν βλέπουμε την ώρα να έχουμε και άλλη ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much for... Σας ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας ε, τις ε, σκέψεις σας ε, σχετικά με <clears throat> τις κινήσεις μας. Ο από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ε, είπατε τι ακριβώς θα πρέπει να αντικατοπτρίζει η νέα κοινή αντίληψη, ότι θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το θεματολόγιο του 2030. Ε, άλλωστε, υπάρχουν ε, τα θέματα ειρήνης, δικαιοσύνης και διακυβέρνησης ε, που θα πρέπει να είναι ένα από τα σημεία κλειδιά που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη νέα κοινή αντίληψη. εξετάζοντας αυτά που λέει το ε, Γερμανικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης όσον αφορά το θέμα της δημοκρατικής διακυβέρνησης μεταξύ άλλων. Βλέπουμε ότι αυτά ευθυγραμμίζονται απολύτως με τις ιδέες του ΕΛΚ. Θα θέλαμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τις, τις πτυχές αυτές και να αντικατοπτρίζονται οι πτυχές αυτές στην έκοινη αντίληψη που φυσικά καλύπτει ε, και πολλά άλλα θέματα όπως είναι η χρηματοδότηση των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και άλλα τέτοια θέματα. Αυτό συνδέεται και με τον ε, ορισμό της ε, επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, κάτι που θα συζητήσουμε αργότερα και με τον Όσα. Και νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στη νέα κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη. Όσον αφορά την συμμετοχή διαφόρων φορέων, ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα, και όχι μόνο στην αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων ε, θεμάτων όπως είναι η ασφάλεια, είναι ένα θέμα στο οποίο συμφωνούμε. Πιστεύουμε ότι οι προτεραιότητες ε, της αναπτυξιακής βοήθειας που στόχο έχουν να γίνουν οι θεσμοί πιο ανοιχτοί και πιο συμμετοχικοί ε, αποτελεί ένα σημείο κλειδί για να πετύχουμε την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτά ήταν κάποια θέματα τα οποία θα ήθελα να επισημάνω σε αυτήν την πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την νέα κοινή αντίληψη. Φυσικά θα προχωρήσουμε βαθύτερα στη συζήτηση αυτή ε, κατά την εκπόνηση της έκθεσής μας. Και προσλέπουμε στο νέο έγγραφο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σαλ Κέρενς. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Χάγενεχ, η οποία μας παρουσίασε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση. Όντως υπογράμμισε τα πιο σημαντικά ζητήματα. Λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση είναι εξή. Τι γίνεται αν δεν συμφωνήσουμε με την Επιτροπή και το Συμβούλιο ώστε να υπάρχει αυτή η συνένεση για την ανάπτυξη. Δεύτερον, τι γίνεται αν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε μαζί τους. Τίποτα, όπως και στην πρώτη περίπτωση. Στη δεύτερη περίπτωση, εκτός αν πάρουμε στα σοβαρά αυτά που αναφέρει το έγγραφο. Και το πρώτο που πρέπει να σημειώσουμε εδώ είναι ότι δεν πήραμε στα σοβαρά το έγγραφο αυτό. Τη δυνατότητα δηλαδή συνομιλίας με το Συμβούλιο. Απουσιάζει πάντα. Υπάρχει κάποιος γύρω από το τραπέζι για να φτάσουμε στο κείμενο και μετά εξαφανίζεται. Όταν λοιπόν διαπιστώσουμε την αποτυχία της χρηματοδότησης, δεν μπορούμε να τηρήσουμε μια βασική αρχή με την οποία συμφωνήσαμε, που είναι η χρηματοδότηση αυτή του 0,7% για αναπτυξιακή βοήθεια μπορούμε να φανταστούμε και μια νέα συνένεση ευρωπαϊκή για την ανάπτυξη που να λέει ότι αν μετά από 15 χρόνια δεν καταφέραμε να πετύχουμε αυτό που υποσχεθήκαμε το 2015, το 2030 ή ένα-δυο χρόνια πριν θα συμφωνήσουμε για μια νέα προθεσμία. Να αναβάλουμε για αργότερα δηλαδή ότι δεν μπορέσαμε να πετύχουμε μέχρι τότε. Η μέθοδος λοιπόν που θα ακολουθήσουμε είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι τα λόγια που λείπουν η θεωρία. Είναι η βούληση να γίνουν όλα αυτά πράξη. Και πώς θα ελεγχθεί η εφαρμογή όλων αυτών που υποσχόμαστε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί ελέγχου. Πρώτος στόχος λοιπόν στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων θα έπρεπε να ήταν ότι αν συμφωνήσουμε πάνω σε κάτι Ας το κάνουμε κιόλα. Και ας έχουμε και τα μέσα να ελέγξουμε κατά πόσο αυτά που υποσχεθήκαμε έγιναν. Ο κατάλογος των αποτυχιών είναι μεγάλος, δυστυχώς. Δεύτερον, πιο υπεύθυνοι, πιο αποφασισμένοι, με περισσότερη συνοχή, περισσότερη καινοτομία και πιο αποφασισμένοι και συγκεκριμένοι στα όσα θα κάνουμε. Τώρα, υπογραμμίσατε και κάτι άλλο που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι πώς θα συνεχίσουμε να εφαρμόσουμε την αρχή της διαφοροποίησης. Είχαμε την επιλογή να πούμε μετά από μια διαπίστωση που ήταν ότι χώρες μεσαίου εισοδήματος μπορούν να παράξουν πλούτο που να πάει στην ανάπτυξη. Και είχα πει 50% των πόρων θα πάνε στις πιο ευάλωτες. Το υπόλοιπο 50% θα είναι ή στις αναδιόμενες ή στις ε, βιομηχανοποιημένες, σε όλες μαζί. Μα τι θα κάνουμε απ' Θα συνεχίσουμε να δίνουμε χρήματα από τη δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια για τους φτωχούς της αναδιόμενης χώρες. Η Επιτροπή έκανε μια επιλογή που τη στήριξε και το Κοινοβούλιο μας και που ήταν να παραιτηθεί από αυτήν τη χρηματοδότηση. Πώς θα ελέγξουμε οι αναδιόμενες χώρες κατά πόσο αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Δηλαδή να μην τρώνε από τα κονδύλια τα οποία έτσι καλλιώς χρειάζονται τόσο πολύ. Η χρηματοδότηση του Trust Fund για την Αφρική, μα Πήγαμε. Ένα σωρό ανακοινώσεις, 12% υλοποιούνται από αυτά που ακούσαμε στην διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρική. Ε, τη διακυβέρνηση ναι και τα άλλα συμφωνώ, αλλά υπάρχει και κάτι που πρέπει να προσθέσουμε. Πέρα από αυτά που σας είπα για τη μεθοδολογία και την εφαρμογή, υπάρχει και το θέμα της περιφερειακής διάστασης, που πιστεύω ότι είναι ζωτική σημασίας πριν συζητούσαμε για τη μετανάστευση, που είναι και ενδοπεριφερειακή. 80% των φτωχών μετακινούνται από τη μία περιφέρεια στην άλλη μέσα σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη. Και εδώ λοιπόν χρειάζεται κάποια απάντηση για να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα και την διακυβέρνηση και σε περιφερειακό επίπεδο. Και έρχομαι στο τελευταίο μου, που είναι ζωτική σημασία. Θα το αντιμετωπίσουμε. Χρηματοδοτική βοήθεια. Πρώτο, τι θα μας προτείνετε ώστε τα χρήματα που κατευθύνονται στην αντιμετώπιση της φτώχειας δεν θα φτάσουν σε αυτούς που αγωνίζονται για την προστασία του κλίματος. Διότι Υπάρχει ζήτημα για το πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά. Ούτε η Επιτροπή, ούτε οι χώρες μέλη δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν μέχρι τώρα για μια σαφή διάκριση των κονδυλίων. Τι θα πάει δηλαδή στην καταπολέμηση της φτώχειας. Αν γίνει αποδεκτός ο ορισμός, δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείτε κάτι διαφορετικό με αυτά τα κονδύλια, γιατί το κάτι διαφορετικό, το κλίμα για παράδειγμα, πρέπει να χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή. Δεύτερον, και αυτό θα συζητηθεί πολύ στο μέλλον, πώς θα χρηματοδοτήσουμε την ενίσχυση της διακυβέρνησης, της ασφάλειας. Γιατί κάθε φορά που γίνεται μια τρομοκρατική ενέργεια, μια επίθεση, θα έχουμε την τάση να χρηματοδοτούμε για την ασφάλεια. Πληροφορίες, υπηρεσίες πληροφοριών, δημόσια τάξη. Αλλά όλα αυτά θα βγαίνουν από κονδύλια που κανονικά θα έπρεπε να πάνε στην ανάπτυξη ή από κάτι άλλο. Ξεκάθαρη η στρατηγική. Πρέπει να καταγραφούν όλες οι ανάγκες και μετά να ρωτήσουμε τις χώρες μέλη αν είναι διατεθειμένες να τα χρηματοδοτήσουν επίσης. Όταν βλέπω τη βούληση των χωρών μελών να παραμείνουν σκλάβοι του 1% του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την δυνατότητα και το Αναπτυξιακό Ταμείο να συμπεριληφθεί σε λίγα χρόνια μέσα στον Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, φοβάμαι ότι όλα αυτά θα γίνουν σε βάρος της αναπτυξιακής πολιτικής. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ένας κατάλογος με όλες τις ανάγκες <coughs> αλλά και με τους κινδύνους. Θα συμφωνούσατε εσείς να φροντίσετε να ακουστεί η φωνή του Κοινοβουλίου. Ένα ε, ζητάμε. Να τηρούν τις υποχρεώσεις τους οι χώρες μέλη, να είναι ε, μετρήσιμα τα όσα κάνουν και να επιδέχονται έλεγχο. Για να γίνει αυτό, η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποκτήσουν εξουσίες. Δηλαδή να έρχονται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσοι άλλο λένε και άλλο κάνουν τελικά αυτή η κοροϊδία όπου ατιμωρητοί ξεφεύγουν όλοι και άλλα υπόσχονται και άλλα κάνουν πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να είναι υπόλογοι, να έρχονται εδώ και να δίνουν λόγο. Αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε σοβαροί με την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Βοήθεια, τότε δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνεται ένα συλλογικό ψέμα όλη αυτή η ιστορία. Με την προηγούμενη Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη έχουμε αρκετές εμπειρίες. Πρέπει να σταματήσει εδώ αυτό το κακό. Μαρία Χόικα. Ευχαριστώ πολύ την ε, κυρία Χακενέσου που ήρθε εδώ στην Επιτροπή μας ε, και που μας παρουσίασε τις θέσεις της. Ε, και ο Σαλκιόρενς αναφέρθηκε στον πιο δεσμευτικό χαρακτήρα ε, θα ήθελα όμως όσον αφορά την ε, πολιτική συνοχή να τονίσω ότι είναι σημαντικό να γίνει σωστή ε, εφαρμογή. Στην εμπορική και γεωργική πολιτική, όταν μιλάμε για τα δικά μας συμφέροντα, ξαφνικά βλέπουμε η πολιτική συνοχή να εξατμίζεται. Τίθεται το θέμα εάν αρκεί η χρηματοδότηση και όταν μιλάμε για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και για το COP21, αλλά παρόμοιο ερώτημα τίθεται για μένα όταν μιλάμε για θέματα ασφάλειας. Ειδικά στις ε, ευάλωτες χώρες ε, τονίζεται η ανάγκη για ασφάλεια, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια αντίφαση όταν ε, μιλάμε για χρηματοδότηση της ασφάλειας από τους πόρους της ανθρωπιστικής βοήθειας. Συμφωνώ απολύτως με τον Σάλ θα πρέπει να δούμε τι θέλουμε να στηρίξουμε και να το χρηματοδοτήσουμε και όχι να αναφέρουμε ένα σωρό θέματα για τα οποία τελικά να μην παρέχουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση. Επίσης, ε, στην ε, κοινή αντίληψη ε, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα αν συμμετάσχει και ο ιδιωτικός τομέας. Θα πρέπει όμως να έχουμε και δεσμευτική ευθύνη του ιδιωτικού τομέα όταν μιλάμε για περιβαλλοντικά πρότυπα, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τέτοια. Αυτές είναι οι γενικές μου παρατηρήσεις. Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η κοινή αντίληψη θα συνεχίσει να χωρίζεται στα δύο, δηλαδή από τη μία να έχουμε τις αρχές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και από την άλλη την ε, κοινοτική πολιτική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και η δεύτερη ερώτηση είναι ο κώδικας δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης για τη συμπληρωματικότητα και το καταμερισμό εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική συνδέεται στενά με την κοινή αντίληψη. Πώς θα επηρεάσει λοιπόν η αναθεώρηση της κοινή αντίληψης ή τον κώδικα δεοντολογίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μαρία. Κάποιες παρατηρήσεις από μένα και κατόπιν θα δώσω το λόγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσες οι προτάσεις σας. Φυσικά συζητάμε και το μέλλον της Συμφωνίας Κοτονού. Θα πρέπει να συνδυάσουμε τα δύο αυτά και φαίνεται να προτείνεται ότι δεν θα πρέπει να έχουμε προνομικές σχέσεις με κάποιες χώρες ε, και να αποκλείουμε κάποιες άλλες, ε, να μην υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, νομίζω ότι αυτό είπατε. Είπατε δηλαδή ότι θα πρέπει να καταργηθεί η συμφωνία του Κοτονού. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω τη θέση σας πάνω σε αυτό. Και θα ήθελα επίσης ε, συγκεκριμένα παραδείγματα χωρών που θεωρείται ότι ε, ε, έπεσαν θύματα διάκρισης. Νομίζω επίσης ότι είναι σημαντικό το θέμα της ασφάλειας, πώς δηλαδή ταιριάζει η αναπτυξιακή πολιτική με την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει μια ευρύτερη πολιτική ασφάλειας. Όσον αφορά τις χώρες μεσαίου εισοδήματος. είπατε ότι θα πρέπει να αποτελούν μέρος της συζήτησης. Μήπως μπορείτε να μας πείτε ποιο πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεων αυτών ε, και οι συνομιλίες μας ε, με τις χώρες μεσαίου εισοδήματος ε, δεν αφορούν μόνο την αναπτυξιακή βοήθεια. Με την Κένια, για παράδειγμα, δεν συζητάμε τόσο πολύ την αναπτυξιακή βοήθεια όσο την εμπορική πρόσβαση και τέτοια. Αν όμως επικεντρωθούμε υπερβολικά στις χώρες μεσαίου εισοδήματος δεν υπάρχει ο κίνδυνος ε, να ξεχάσουμε το θέμα της στόχιας, ε, διότι η στόχοι της χιλιετίας είχαν να κάνουν με την εκρήρωση της στόχιας. Ε. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης είναι πολύ ευρύτεροι και ε, ε, ασχολούμαστε με κάποιες από τις χώρες που θα επηρεαστούν περισσότερο από την αλλαγή του κλίματος, ε, κάποιες χώρες σε νησιά. Πώς λοιπόν θεωρείτε Θεωρείται μάλλον ότι θα είναι σημαντικό στην νέα κοινή αντίληψη να επικεντρωθούμε πάλι στη φτώχεια. Επίσης είχαμε την ε, πρόταση των συντονιστών ε, να έχουμε κάποιες έρευνες ε, σχετικά με το Πώ έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να ξέρω τι έχει αλλάξει από το 2005 μέχρι το 2015 στην αναπτυξιακή πολιτική. Είδαμε να υπάρχει περισσότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Είδαμε πιο συνεκτική πολιτική στην πράξη. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον, ε, διότι ε, είναι πολύ ωραίε οι θεωρίε περί αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά ε, το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη. Ο κόσμος νιώθει την αλλαγή ή έχουμε, διάφορες, ή έχουμε διάφορα ημιτελή προγράμματα τα οποία ε, κλείνουν ε, χωρίς να έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Θα δώσω τον λόγο στον Κάσπαρ Φοντίνη από την Γενική Διεύθυνση Ντεύκο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να ακούσω την ε, συζήτηση αυτή, η οποία νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για μας. Νομίζω ότι Ακριβώς αυτό θα πρέπει να κάνουμε κατά την εκπόνηση της κοινή αντίληψης. Ε, να έχουμε μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με εσά και με διάφορους άλλους παράγοντες. Πέρα από αυτό, επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις που νομίζω ότι θα είναι χρήσιμες για τη συζήτηση αυτή. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι, αν εξετάσουμε την αντίδραση στην, στο θεματολόγιο του 2020 και τις προσπάθειες επικαιροποίησης ε, της ε, κοινή αντίληψης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπτυξιακή πολιτική, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αποτελεί μέρος της αντιμετώπισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης του θεματολογίου για το 2050 και είναι σημαντικό να δούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα αντιμετωπίσει ε, τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές του θεματολογίου αυτού. Θα πρέπει να δείξουμε λοιπόν ότι κάνουμε πράγματα και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά θέματα κλειδιά τα οποία θα ε, αντιμετωπίσουμε σε άλλα έγγραφα τα οποία δεν σχετίζονται με την κοινή αντίληψη. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να υπάρχει συνεκτικότητα και να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλέ πτυχέ στο θέμα αυτό που δεν αντικατοπτρίζονται όλε στην κοινή αντίληψη. Δεύτερον, όταν μιλάμε για την επικαιροποίηση τη κοινή αντίληψη, ε, σημαντικό είναι να ληφθεί υπόψη το θεματολόγιο 2030. Το προηγούμενο θεματολόγιο βασιζόταν ε, στι στόχου τη χιλιετία. Ε, τώρα έχουμε κάποιε καινοτομίε οι οποίε θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται πλήρω στη νέα κοινή αντίληψη. Αυτή όμω δεν είναι η μόνη αλλαγή στο διεθνέ σκηνικό. Είχαμε και τη διάσκεψη του Παρισιού και άλλες ε, που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη νέα κοινή αντίληψη. Επιπλέον θα πρέπει να σκεφτούμε όλες τις τάσεις που αναφέρονται εδώ και να προσπαθήσουμε να τις εσωματώσουμε. Κάποιες από αυτές ε, ήδη αντικατοπτρίζονται στο θεματολόγιο 2030. Θα πρέπει όμως ε, να γνωρίζουμε ότι αν θέλουμε να είμαστε επίκαιροι θα πρέπει στην αντιμετώπιση μας να συμπεριλάβουμε όλες τις τάσεις που βλέπουμε στον κόσμο και στην οικονομία. Τρίτη παρατήρηση. Θέλουμε όλα αυτά να γίνουν με μια πολύ ισχυρή διαδικασία διαβούλευσης με εσάς, με τα κράτη-μέλη, με την κοινωνία των πολιτών, με τον ιδιωτικό τομέα. Θα εργαστούμε πάνω στο θέμα αυτό, θα ξεκινήσουμε εξωτερική διαβούλευση πολύ σύντομα. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μα, θα πρέπει να το κάνουμε μαζί σα και θα πρέπει να έχουμε μια πολύ ευρία διαβούλευση. Όσον αφορά τα θέματα που αναφέρθηκαν εδώ, ε, σχετικά με το περιεχόμενο τη νέα κοινή αντίληψη, Φυσικά είναι πολύ νωρί ακόμα να πούμε ποιο θα είναι το τελικό περιεχόμενο. Νομίζω όμω ότι πολλά από τα θέματα που αναφέρθηκαν εδώ θα είναι κλειδιά στη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι στο θεματολόγιο του 2030 υπάρχει η βούληση να συνδυαστούν θέματα βιωσιμότητας και μείωσης της στόχιας. Και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να το μεταδώσουμε αυτό στον κόσμο, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρες και τις αναπτυσσόμενες χώρες να πετύχουν τους δικούς τους στόχους και τις δεσμεύσεις τους στη, στο θεματολόγιο και πώς θα συνδυάσουν τις διάφορες στοιχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Όσον αφορά την, ε, τις εξελίξεις, όσον αφορά τη φτώχεια. Βλέπουμε ότι η φτώχεια έχουμε κυρίως σε χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις ή χώρες ασταθείς. Ε, εδώ δεν βλέπουμε να υπάρχει πρόοδο όσον αφορά του στόχου τη ε, χιλιετία και θα πρέπει να δούμε πώ θα μπορούμε να επικεντρωθούμε στο θέμα αυτό. Θα πρέπει δηλαδή να συνδέσουμε τα θέματα αυτά με ε, την ε, πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας και άλλε πολιτικέ. Έχουμε ακριβώ τη δυνατότητα να ενισχύσουμε σε διαφορετικά επίπεδα, το οποίο είναι πλέον έκτημα. Από την άλλη πλευρά έχουμε αναπτυσσόμενες χώρες που αναπτύσσονται και και ε, με κάποιες από τις χώρες αυτές θα προχωρήσουμε σε διμερή συνεργασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν πια προβλήματα, αλλά θα πρέπει να δούμε τι είδους συνεργασία θα βοηθήσει τις χώρες αυτές. Τέλος, κάτι που δεν αναφέρθηκε, το οποίο όμως νομίζω ότι είναι σημαντικό, είναι το θέμα των ανισοτήτων. Μεταξύ άλλων, μεταξύ των δύο φύλων. Τα θέματα αυτά τονίζονται ιδιαίτερα στο θεματολόγιο 2030 και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εισάγουμε τα θέματα αυτά στην κοινή μας αντίληψη. Και για να κλείσω τη σύντομη παρέμβασή μου, νομίζω θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά τους τρόπους εφαρμογής όλων αυτών. Η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα για κάποιε χώρε Υπάρχουν σαφείς τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα πρέπει Όμω επίσης να κινητοποιήσουμε και άλλες πηγές χρηματοδότηση, κάτι το οποίο θα πρέπει να σκεφτούμε. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι να υπάρχει συνεκτικότητα στην πολιτική μας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξετάζουμε πώς μπορούμε αυτή η συνεκτικότητα στις πολιτικές μας να αποτελέσει πραγματικότητα και πώς θα μπορεί να αντικατοπτρίζεται αυτή στην κοινή αντίληψή μας για ε, ανάπτυξη. Ευχαριστούμε. Πολύ χρήσιμο διότι λέτε ότι η πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καθορίσει στόχους για μετά το 2030 είναι κάτι που θα γίνει σύντομα. Καλό θα ήταν αν μπορείτε να ενημερώσετε και τη γραμματεία μα, να στείλουμε εμεί κάποιο συνεργάτη, ώστε να έχουμε μια επισκόπηση του τι θα συμβεί και τι θα συζητηθεί. Είναι σημαντικό για την κοινή αντίληψη και το πώ θα δημορφωθεί, αν γίνονται και κάποια πράγματα ταυτόχρονα. Από ό,τι κατάλαβα, λοιπόν, θα πάρουμε την ανακοίνωση για το τι θα γίνει μετά το 2030 για την εξωτερική δράση, αλλά αυτό θα αντικατασταθεί από την κοινή αντίληψη, είχαμε καταλάβει ω τώρα, τώρα μα λέτε κάτι διαφορετικό. Να είμαστε σαφεί, εάν γίνεται. Ή τέλο πάντων να τα δούμε στη συνεδρίε των συντονιστών. Να υπάρχει σαφήνεια στο τι θα κάνει η Επιτροπή. Θα μα εξυπηρετήσει αυτό για το μέλλον. Να ξαναδώσω το λόγο στην Κριστίν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι αν είμαστε επίκαιροι ή όχι. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση έχει αλλάξει πολύ από το 2005. Έχουμε πλέον εκπρόσωπο για τι ε, εξωτερικέ μα σχέσει που βρίσκεται με το ένα πόδι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με το άλλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό δυσκολεύει βεβαίω και την κυλιόμενη Προεδρία του Συμβουλίου, την αναλωσόμενη Προεδρία, να έρθει να τοποθετηθεί για τα θέματα αυτά. Η ανθρωπιστική βοήθεια, ναι, σχολιάζεται, αλλά όχι αναπτυξιακή. Νομίζω λοιπόν ότι η επίκριση που εξέφρασα προς τα κατημέλη και το Συμβουλίο είναι ότι θα πρέπει να βρουν στο επίπεδο του Συμβουλίου μια απάντηση για το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Προεδρία της. Εφόσον εκείνοι θα έχουν την τελευταία κουβέντα που θα είναι και πιο σημαντική για να πούν στην ε, πολιτική και τον προγραμματισμό της ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια απάντηση. Ναι. Έτσι φαίνεται, γιατί οι υπουργοί φαίνεται να συναντιούνται και να μην μιλάνε για ανάπτυξη. Αν πάει όμω κανεί στο άτυπο συμβούλιο, βλέπουμε Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να προεδρεύει πολλέ φορέ το ίδιο το Συμβούλιο και να καθοδηγεί τι συζητήσει. Και τελικά δεν συμβαίνει αυτό στι επίσημε καταστάσει. Είναι μια περίεργη σύμβαση αυτή. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έρχεται και να λέει αυτά που θέλει να πει, όμω όντω τα κράτη-μέλη πιέζουν. Πιέζουν και πολλέ φορέ απλώ συντονίζει η εναλλασσόμενη Προεδρία. Τα σημειώνουν οι συνεργάτε μα Κριστίνα, λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους για τα τόσο ενδιαφέροντα σχόλια και ερωτήσεις. Θα σταθώ επιλεκτικά σε κάποια στοιχεία και θα απαντήσω σε ορισμένες ερωτήσεις. Και θα πάω ίσως ανάποδα, γι' αυτό θα ξεκινήσω με τις δικές σας ερωτήσεις. Αυτό που σχολιάσατε για την συνεργασία με τις ε, χώρες μέσω εισοδήματο και το κατά πόσον μπορούμε να επικεντρωθούμε σε αυτά και για το εάν θα παραμελήσουμε τις χώρες ε, τις λιγότερο αναπτυγμένες ή τις αναπτυσσόμενες. Δεν είναι κοντρό να επικεντρωθούμε μόνο στις χώρες μέσω εισοδήματος, απλώς η βοήθεια στις χώρες ανώτερου μέσω εισοδήματος βλέπουμε να επικεντρωθουμε μονο στις χωρες μεσω απλως η βοηθεια στις χωρες ανωτερου μεσοσοδηματος βλεπουμε να μειωνεται και να περικόπτεται, οπότε έχει παραμείνει ένα κάποιο κενό ένα χάσμα το οποίο καλό θέλει να καλυφθεί για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε συνεργασία με τις χώρες αυτές και να αντιμετωπίσουμε κοινέ προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε να δούμε τα εργαλεία μας για τα κοινοφελή αγαθά και το κατά πόσο η ανεπτυξιακή βοήθεια μπορεί να αξιοποιηθεί για να συνεργαστούμε με τι χώρε αυτέ. Βεβαίω, ο μεγαλύτερο όγκο τη βοήθεια πρέπει να πάει προ τι χώρε χαμηλού εισόδηματο και αυτέ που είναι λιγότερο αναπτυγμένε. Μετά για τι χώρε ΑΚΕ έγιναν κάποια σχόλια. Αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται παράλληλα ε, και είναι πολύ σημαντική. Σίγουρα χρειάζονται εδώ ριζικέ μεταρρυθμίσει των σχέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τι χώρε αυτέ. Αλλά μεταρρύθμιση μπορεί να σημαίνει ότι πτυχέ που έχουν καθοριστεί από πολύ παλιά και ήταν θετικέ ω τώρα στι σχέσει μα, μπορεί να χρησιμεύσουν και σε άλλα τμήματα των σχέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τι χώρε αυτέ. Όπω ο προσανατολισμό του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου προς συγκεκριμένους στόχους. Αυτό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και από άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία και μηχανισμούς. Η ερώτηση του κυρίου Χόιμπουχ για τον ευρωπαϊκό συντονισμό εντός της Ευρωπαϊκής Κοινής Αντίληψης. και τα εργασιακά Νομίζω ότι υπάρχει εδώ ένα κοινό προγραμματισμό και θα πρέπει και μια αντίληψη να αποστείλει ένα στεναρό μήνυμα για την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών κλάδων και τομέων. Αυτό θα είναι μια σημαντική παράμετρο τη νέα κοινή αντίληψη. Και μια τελευταία παρατήρηση, ίσω, για να επανέλθω σε μια από τι δικέ σα ερωτήσει. Τι γίνεται. Συμφωνώ η συζήτηση αυτή είναι φιλόδοξη. Γεμάτη δυσκολίες. Τι θα γίνει αν δεν καταλήξει σε συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοινή αντίληψη, αν δεν είναι αρκετά φιλόδοξη αυτή η νέα κοινή αντίληψη. Σημαντικό το θέμα. Υπάρχουν πολύ ψηλές προσδοκίες από τις χώρες εταίρους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταλήξει σε μια φιλόδοξη συμφωνία μεταξύ των διαφορών θεσμών. Υπάρχει ένα ζήτημα αξιοπιστία όμω. Είναι και αυτό σαφέ. Οπότε παρόλο που αναγνωρίζω ότι θα είναι δυσκερή οι συζητήσει, νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση στι συζητήσει τη να αποστείλει ένα χειρομήνυμα Ότι είναι αφοσιωμένη στο να έχει μια εντατική κοινή προσπάθεια για την αναπτυξιακή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Αυτή ήταν η πρώτη μια ολόκληρη σειρά από συζητήσει και ανταλλαγέ απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για την κοινή αντίληψη, το consensus όπω λέγεται. Μα δώσατε πάρα πολύ υλικό για σκέψη και σα ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Να θυμίσω σε όλου ότι θα ψηφίσουμε στι τρει οπότε παρακαλώ φέρτε τι κάρτε σα. Και θα σα δω το απόγευμα.